ζήτημα αυτό στη νομική επιτροπή που είναι αρμόδια. Επόμενο θέμα. Έχω λάβει αιτήματα τροποποίησης από πλευράς του Λαϊκού Κόμματος για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Θα βρείτε την αντίστοιχη λίστα στο ο πρακτικό της παρούς συνεδρίασης και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ο κατάλογος αυτός ε, γκριθής. Επίσης θέλω